Τώρα έχουμε μία σύντομη παρουσίαση της έκθεσης Βαλέαν για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους στην επικράτεια των κρατών μελών. Το λόγο έχει ο συγγητής για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε. Από τα βασικά δικαιώματα των πολιτών ένα που μας ενώνει όλους είναι το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Αυτό το προβλέπουν οι συνθήκες και το εφαρμόζει η Οδηγία 38 του 2004 που εκφράζει και τα δικαιώματα και τους περιορισμούς που πρέπει να εφαρμόζουν οι πολίτες, τα υποχρεώσεις, για να κινούνται ελεύθερα στο έδαφος της Ένωσης. Το 2006 πάνω από 8 εκατομμύρια πολίτες άσκησαν το δικαίωμα αυτό να κατοικήσουν σε μια τρίτη χώρα και να ταξιδεύσουν. Ω εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αξιολόγηση τη οδηγία αυτή, πρέπει να σα πω ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή άσκηση του δικαιώματο αυτή τη ελεύθερη διακίνηση των πολιτών υπονομεύεται σοβαρά από τα κράτη-μέλη κατά παραβίαση των συνθήκων και της οδηγίας. Πρώτον, για τη μεταφορά στα στο δίκαιο των κρατών μελών. Δεν έγινε πλήρως. Σε δύο μελέτες της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου ταυτίστηκαν τα προβλήματα. Πρόκειται για παραβίαση δικαιωμάτων των πολιτών και αυτό φαίνεται, το δείχνω στην έκθεσή μου. Τίθενται πολλά δικαιολόγητα, δικαιολόγητη γραφειοκρατική φραγμή, ιδίω για οφείλονται κυρίως σε διαδικαστικές καθυστερήσεις και περιορίζεται η κυκλοφορία ορισμένων εταίρων γνωστών από τον νόμο που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν όπως θέλουν. Επίσης, αγνοείται η αρχή της αναλογικότητας και έτσι ορισμένοι πολίτες δεν τυχαίνουν ίσης μεταχείρισης με άλλους. Αντίθετα με αυτά που προβλέπει η οδηγία. Έπειτα. Συμφωνώ ότι είναι σοβαρά τα προβλήματα, αλλά το άρθρο 38 της οδηγίας ήδη προβλέπει τη δυνατότητα των χωρών μελών να καταπολεμήσουν καταχρήσεις όπως τους γάμους ευκαιρίας. Επίσης, συνεργάστηκα επικοδομητικά με Εθνικά Κοινοβούλια την Κομισιόν καθώς και την κυρία Μόνικα Φρασόνη που ήταν η συγγήτρια της Νομικής Επιτροπής. Η έκθεσή μου επίσης ζητάει ορισμένα μέτρα και ένα από τα σημαντικότερα είναι η δημιουργία από την Κομισιόν συγκεκριμένων κατευθυντηρίων γραμμών για τη μεταφορά της οδηγίας. Με τη διασφάλιση βέβαια του δικαιώματο των κρατών μελών να απολαμβάνουν τις ασφαλείας τους. Η ακατάλληλη μη ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών αποτελεί παραβίαση και πρέπει τελικά να υπάρξει αναθεώρηση της, ε, πολλα, πλη, της ε, πλημελούς αυτής μεταφοράς στα, εθνικό, στα εθνικά δίκαια. Επίσης, η Κομισιόν δεν πρέπει να διστάσει να προσφύγει κατά χωρών μελών που δεν εφαρμόζουν την οδηγία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν και να μεταφέρουν σωστά την οδηγία για να λυθούν τα προβλήματα και να μην προσπαθήσουν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους για να νερώσουν την οδηγία, να αποδυναμώσουν την οδηγία. Εμείς είμαστε κατά μια τέτοια αποδυνάμωσης και ευτυχώς και οι Κομισιόν επίσης. Καιρός είναι και τα τρία όργανα να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία όχι μόνο των αγαθών και των κεφαλαίων αλλά και των πολιτών γιατί χωρίς την ελεύθερη κυκλοφορία δεν υπάρχει Ευρώπη. Τέλος, κατέθεσα μία τροποποιημένη προφορική τροπολογία για να μην έχουν καμία δικαιολογία ορισμένοι που αρνούνται την ε, ίση μεταχείριση για λόγους ομοφοβίας και άλλους παρόμοιους που δεν τολμούν να τους πούν καθαρά. Στην πληροφορία θα δούμε ποιος είναι πράγματι υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας και ποιος όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η απάντηση της Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά κυρία εισηγήτρια, εσάς προσωπικά, για μια αξιοπρόσεκτη πολύ καλή έκθεση. Και θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή επικοδομητική συνεργασία σε ένα πάρα πολύ ακαθόδες θέμα. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων είναι μία από τις ουσιοδέστερες ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Εσωτερική Αγορά η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων είναι αυτό το οποίο δημιουργεί την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ως θεμέλιο και τεκμηριώνει και θεμελιώνει την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και είναι σαφές ότι ελλείψεις ή μειονεκτήματα όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε αυτό το τομέα αποτελούν πράγματι μια παραβίαση έναντι των πιο θεμελιωδών αρχών που αφορούν και δημιουργούν τα θεμέλια της Ευρώπης και εδώ πρόκειται για ένα κέριο σημαντικότατο στοιχείο και γι' αυτό χαιρετίζω για αυτούς τους λόγους την έκθεση αυτή που <clears throat> σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2008 για την ε, εφαρμογή της ε, σχετικής οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι ουσιαστικά ότι πρακτικά όλα τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμπίπτουν με τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έλεγα ότι τώρα έχουμε μια πλήρη εικόνα, πλήρη εικόνα της υλοποίησης και εφαρμογής της οδηγίας στα κράτη-μέλη, επιτόπου δηλαδή, χειροπιαστά. Και ήρθε τώρα ο χρόνος να δράσουμε αποτελεσματικά. Στην έκθεση αναφέρεται και τονίζεται και δίκαια αυτό ότι η αρμοδιότητα για την ορθή και δέουσα εφαρμογή αυτής της οδηγίας η αρμοδιότητα είναι των κρατών μελών αποκλειστικά. Όμως, ωστόσο, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς να δραστηριοποιείται. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου να επεξηγήσω πού ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε αυτά τα πλαίσια βλέπει να υπάρχουν άμεσες προτεραιότητες για αυτήν για να δραστηριοποιείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί μεγάλη σημασία η οδηγία πλήρως και με ορθό τρόπο να εφαρμόζεται. Είναι μία από τις προτεραιότητες αυτή για μας. Στην 25η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, την εφαρμογή και τον έλεγχο του κοινοτικού δικαίου 2009 λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίζει ότι η κατεύθυνση αυτή, η οδηγία αυτή ε, πλήρως και με ορθό τρόπο θα εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ με τα κράτη-μέλη με προσπάθειες που έγιναν ώστε η πολλαπλά ελληματική ή με ε, ελλείψεις εφαρμογή να αντιμετωπιστεί σωστά. Αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικά αποτελέσματα από αυτή την προσπάθεια και συνεργασία δεν θα διστάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα να προσφύγει στο ΔΕΚ λόγω παραβίας, παράβαση, επιπαραβάση εις βάρος των κρατών μελών που δεν θα ε, τηρούν ε, τις ορθές διαδικασίες. Στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έναντι των κρατών μελών και έναντι των πολιτών να διαχέει και να διαθέτει αναγκαίες χρήσιμες πληροφορίες ώστε κατευθυντήρες για παράδειγμα ε, γραμμές να καταρτίζονται για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας σε συγκεκριμένους ίσως προβληματικούς τομείς. Για παράδειγμα, στο θέμα της ε, του εντοπισμού και καταπολέμησης ε, καταχρήσεων, περιπτώσεων κατάχρησης. Στην έκθεση αυτή αναγνωρίζεται ότι εδώ δημιουργείται, υπάρχει ένα επίπεδο ε, που δημιουργεί δυσκολίες. Εδώ θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το επίπεδο να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη ώστε να εντοπίζονται και να καθορίζονται δυσκολίες και θέματα ερμηνείας της εφαρμογής αυτής της οδηγίας να αποσαφηνίζονται. Πρέπει ωστόσο να πω Ευρωβουλευτά ότι την τροπολογία 23 δεν μπορεί να την δεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην πρόταση αυτή τι γίνεται προβλέπεται ότι ομάδες πραγματογνωμόνων θα κάνουν επισκέψεις, αποστολές επί τόπου και με αυτές τις αποστολές θα υπάρχει ένα σύστημα αμοιβαίας αξιολόγησης το οποίο θα εισαχθεί και θα λειτουργήσει. Πρέπει όμως εδώ να επισημάνω ότι τέτοιου είδους αμοιβαίοι έλεγχοι και μέσα σε ένα αμοιβαίο πλαίσιο, μέσα τον τρίτο πυλώνα εντάσσονται και πρέπει εδώ να το δούμε αυτό και όσον αφορά λύσεις και παραδόσεις των κρατών μελών για ε, επίλυση προβλημάτων αυτό σημαίνει ότι η πρόσθετη αξία που θα πρέπει να δημιουργείται από τέτοιους ελέγχους πιθανότατα θα είναι περιορισμένη διότι καθότι γνωρίζετε τα κράτη-μέλη έχουν την επιλογή της μορφής του τύπου και των μέσων για την υλοποίηση και εφαρμογή μιας τέτοιας οδηγίας. Εκεί να επιλέγουν. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διάθεση πληροφοριών για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα. Μια επικαιροποιημένη ε, ε, πρόταση θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή. Επίσης θα ζητήσει από τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τα υποστηρίξει να καταλήξει σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών ε, σε σχέση με τα δικαιώματά τους και σε σχέση με το πώς έχουν τα πράγματα για αυτή την οδηγία. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ε, περισσότερες προτάσεις που έχει υποβάλει η Ευρωβουλή είναι πρόθυμη να τις ακολουθήσει. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωβουλή για την υποστήριξή της και τη συνεργασία της για την διασφάλιση ότι αυτή η σημαντική οδηγία θα μπορέσει σωστά να εφαρμόζεται και μια οδηγία βέβαια όπου πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη σωστή δηλαδή εφαρμογή μιας των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα ερχόμαστε στην σύντομη παρουσίαση της εξέσεως της κυρίας Ρής για τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεφτά. Ευχαριστώ. Δεν είμαι η πρώτη και προφανώς δεν θα είμαι και η τελευταία η